Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Λοιπόν, Continuamos con el punto 10. Συνεχίζουμε με το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση εκφόρτωσης. Γνωρίζετε το ιστορικό αυτής της πρότασης Φτάσαμε σε μια κρίσιμη πλέον στιγμή για προφανείς λόγους και λόγω πίεσης χρόνου. Φτάνουμε στο τέλος της θητείας μας, ο χρόνος πιέζει, κάτι που θα χαρακτηρίσει γενικότερα το φάκελο αυτό. Αυτό γενικά. Τώρα, ειδικότερα πώς ε, εγώ χειρίστηκα αυτή την έκθεση Όπως θα ξέρετε, έγινε μια πρώτη συνάντηση εργασίας για να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, δεδομένου ότι πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα. Υπάρχουν όμως και άλλες αποφάσεις, τις οποίες η Κομισιόν της ενέταξε σε ένα πλαίσιο τεχνικών μέτρων και οι οποίες ε, δεν είναι εξίσου πολύ περισσότερο που ενδεχομένως ε, δεν είναι και ο κατάλληλος τρόπος ε, ε, να ληφθούν. Δεν θέλουμε να δώσουμε μια λευκή επιταγή στην Κομισιόν με αφορμή το ότι πιέζει ο χρόνος. Στη συνάντηση αυτή, στην πρώτη αυτή συνάντηση, ακούσαμε πιο πολύ την Κομισιόν, δεν προχωρήσαμε πάρα πολύ. Και εγώ πρότεινα να χωρίσουμε το θέμα. Αφενός αυτά τα οποία θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2015, πελαγικά ήδη δηλαδή, και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία να τα δούμε πιο προσεκτικά, πιο ήρεμα και αυτά τα δεύτερα να τα αφήσουμε για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Η ομάδα εργασία να ασχοληθεί μόνο με το πρώτο κομμάτι, τα πελαγικά. Τώρα, εμβαθύνοντα, βλέπουμε σιγά σιγά ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τα ξεχωρίσουμε. Ούτε και το πρώτο κομμάτι, τα πελαγικά ήδη είναι τόσο εύκολο να το ρυθμίσουμε μέχρι τον Απρίλιο. Αυτή είναι η γενική εντύπωση. Σήμερα τι θα κάνουμε. Πρώτον, η Κομισιόν θα μας παρουσιάσει την πρότασή της. Λεπτομερώς. Και μετά θα σας δώσω το λόγο να μιλήσετε για το θέμα αυτό γενικότερα. Όχι να μην περιοριστούμε μόνο στην πρόταση Κομισιόν δηλαδή. Να μου μιλήσετε και για τα διαδικαστικά, να δούμε πώς θα βρούμε μια λύση γνωρίζοντας την πίεση του χρόνου και γνωρίζοντας ότι η χρονική πίεση δεν μπορεί να αποτελέσει τον μόνο παράγοντα που θα, αποφασίσει, θα επηρεάσει τις αποφάσεις μας για το μέλλον. Αν δεν έχετε να πείτε κάτι αυτή τη στιγμή, να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Thank you very much, Chair, and good afternoon to... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρουσιάσατε σε κάποιο βαθμό το, ε, το ιστορικό. Να σας πω όμως και εγώ μερικά πράγματα. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε μια ε, νομική ασφάλεια, ευκρίνεια για την καλύτερα, έτσι ώστε όταν τα μέτρα αυτά τεθούν σε εφαρμογή από 1η του 2015 να μην υπάρχουν πλέον ε, νομικές ασάφειες. Έχουμε διάφορα τεχνικά μέτρα αλλά και μέτρα προκύπτουν από τον ε, κανονισμό ελέγχου ε, μέτρα τα οποία αντιβαίνουν με τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης που προκύπτουν από την νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Χρειάζεται αυτές τις νομικές ασυνέπειες οι ασυμβατότητες ε, να τις αντιμετωπίσουμε προς όφελος τόσο των αλλιών όσο και των ελεγκτών των, και των εθνικών αρχών. Θα ήταν καταστροφικό ε, και πολύ δύσκολο άλλωστε να, να αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί σωστά η υποχρέωση εκφόρτωσης αν, για παράδειγμα, οι αλληλείς δεν καταλαβαίνουν τι θα πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το καθήκον τους, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς κατόπιν της ε, ολοκλήρωσης κατά κάποιο τρόπο της κοινή αγροτικής πολιτικής αρχίσαμε όσο πιο γρήγορα γινόταν ε, να επεξεργαζόμαστε αυτές τις προτάσεις. Τις υποβάλαμε τώρα όχι για να πιέσουμε υπερβολικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Απλά ο χρόνο πιέζει έτσι κι αλλιώ. Η κοινή αλληλευτική πολιτική ήταν πλέον έτοιμη στο τέλος του προηγούμενου χρόνου και έτσι μόνο είχαμε τη νομική βάση για να υποβάλουμε αυτές τις προτάσεις πρώτη φάση της υποχρέωσης εκφόρτωσης αρχίζει να ισχύει από 1η 2015. Έχουμε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο δηλαδή. Ο κανονισμός αυτός εξετάζει αφενός τα τεχνικά μέτρα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο επανεξετάζουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και προκειμένου να δούμε αν ε, αντιβαίνουν με την υποχρέωση εκφόρτωσης και δεύτερον, αφετέρου, τα μέτρα ελέγχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα μεγέθη, ε, έτσι ώστε ε, να αποφύγουμε τις παράνομες απορρίψεις ε, και ε, να διαθέτουμε το απαραίτητο σύστημα ελέγχου γι' αυτό. Όλα αυτά είναι μια συνολική ε, διαδικασία και έχουμε ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση τόσο για το πρώτο στάδιο όσο και για τα επόμενα στάδια της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Οι διορθώσεις νομοτεχνικά θα αρχίζουν να ισχύουν ε, στο μέτρο που αρχίζουν να ισχύουν και υποχρέωσεις, υποχρέωσεις εκφόρτωσης. Δηλαδή, οι διορθώσεις δεν θα τεθούν σε εφαρμογή όλες μαζί. Θα υπάρξει ένα πρώτο κύμα 1η Ιανουαρίου 2015, ένα δεύτερο κύμα την 1η 2016 κλπ. κλπ. Αυτά για να είμαστε λογικά συνεπείς στην προσέγγιση μας. Διότι καταλαβαίνουμε ότι ε, σας ζητάμε να εξετάσετε αυτή την πρόταση παράλληλα με την όλη διαδικασία αναμόρφωσης των τεχνικών μέτρων υπό το φως της νέας κοινής αλληλευτικής πολιτικής. η οποία και προβλέπει μια ε, περιφερειακή, ε, μια περιφερειοποιημένη προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε ό,τι χρειάζεται να προσαρμοστεί αυτή τη στιγμή, χωρίς να, να αγγίζουμε οτιδήποτε άλλο, διότι αν το κάναμε ε, θα εμπλεκόμασταν ε, στην ε, διαδικασία διαβούλευση που έχει ήδη ξεκινήσει, η οποία θα οδηγήσει την Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις για την προσαρμογή της ουσίας των τεχνικών μέτρων. Αυτό θα γίνει, ελπίζω, πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί θέλει πραγματικά πολλή δουλειά. Για λόγους πληρότητας, να υπογραμμίσω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας, διότι υπάρχουν τεχνικά μέτρα και στους κανονισμούς της Κομισιόν. Και αυτά τα τεχνικά μέτρα θα ευθυγραμμιστούν με τη νέα πραγματικότητα. Αυτό θα γίνει παράλληλα και βέβαια προφανώς κάθε φορά πριν τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο, η επόμενη φάση ε, υλοποίηση τη υποχρέωση εκφόρτωση. Τώρα, ποιε είναι οι αλλαγέ που προτείνουμε. Θέλουμε να τροποποιήσουμε έξι κανονισμού. Πέντε είναι τεχνικά μέτρα και ο έκτος είναι ο κανονισμό ελέγχου. Και να καταργήσουμε έναν, ε, την ε, βιομηχανική αλία Ρέγκας, που πλέον είναι περιττός. Η λογική των προτάσεων είναι αντί να ε, ρυθμίζουμε τις εκφορτώσεις, να ρυθμίζουμε τις αλλιεύσεις. Δεν είναι έκπληξη αυτή για σας. Για τα τεχνικά μέτρα, η ουσία ε, είναι τρία πράγματα. Ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης, ε, κανόνες σύνθεσης και παραλίευματα ελάχιστα μεγέθη, στην πραγματικότητα είναι αλλάζουμε το όνομα. Στην παρούσα νομοθεσία τα μεγέθη εκφόρτωσης τα αποκαλούμε με διαφορετικούς τρόπους, θα το ενοποιήσουμε. Δεύτερον, σε ό,τι τα μεγέθη δεν αλλάζουν ως αποτέλεσμα αυτής της πρότασης, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε, να σκεφτούμε και την αλλαγή των ίδιων των μεγεθών ε, τη στιγμή που θα χρειαστεί να υποβάλουμε ε, την τις προτάσεις για την αλλαγή των κανονισμών στην ουσία τους. Και οι αλλαγές είναι σταδιακές, όπως σας είπα και προηγουμένως. Για κάθε μία από τις... Ε, ε για ένα από τους διαφορετικούς ε, κλάδους ε, αλλιευμάτων μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. μετά, σύνθεση των αλλιευμάτων ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα αλλιεύματα εκφορτώνονται και συγκρίνονται με τις ε, ποσοστώσεις. Αυτό πώς θα γίνει, κατά βάση με εξαιρέσεις ε, στον σημερινό κανονισμό σύνθεσης. Αν λοιπόν ένας αλίας ανακαλύψει τα δίκτυα του ε, κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλέπονται ή προβλέπεται από τους παλιούς ε, κανόνες, ε, δεν χρειάζεται να ακολουθεί τους παλιούς κανόνες. Δεν αφαιρούμε κάτι για να μην δημιουργήσουμε νομικό κενό μέχρι να αποκτήσουμε τους καινούριου κανόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι διατάξει παρεπιπτών των αλλιευμάτων, ακολουθούμε την ίδια περιπολογική, Δεν αλλάζουμε τα ποσοστά, τα, τις προθεσμίες και όλα αυτά που προβλέπονται από τους κανόνες ε, παραλιευμάτων. Αυτό θα γίνει σε ένα επόμενο στάδιο. στο στάδιο της αναθεώρησης των τεχνικών κανόνων. Τι ό,τι φορά τον έλεγχο, με δύο λόγια αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε επαρκή τεκμηρίωση των ελευμάτων, να καταγράφονται και να αναφέρονται και να συμπεριλαμβάνουμε και τα λεύματα κάτω των ελάχιστων ορίων. Όπως ξέρετε ε, δεν ε, μετράνε τις ποσότητες αλλά θα πρέπει να καταγράφονται. Υπάρχει και ένας ε, αριθμός κανόνων για ε, την ε, εξαποστάσεως ηλεκτρονική παρακολούθηση. Δεύτερον, έχουμε κανόνες για την πρόληψη της αλίευσης μικρών μεγεθών για ανθρώπινη κατανάλωση κανόνες για το πώς θα πρέπει να διατηρούνται στο σκάφος για να, καταμε... για να καταμετρώνται ξεχωριστά. Και τέλος, στην αποτροπή. Ε, περιλαμβάνουμε ε, τις απορρίψεις στις ε, βασικές ε, ε, παραβάσεις του, κανόνα, του κανονισμού. Είπατε ότι πρέπει, ο πρόεδρος μάλλον είπε ότι θέλει να δούμε τι είναι ποιον και τι δεν είναι. Για μας το σημαντικό είναι οποιαδήποτε στιγμή από τώρα μέχρι την τελευταία φάση της εισαγωγής της υποχρέωσης εκφόρτωσης να μην υπάρχουν νομικές ασυμβατότητες διότι αν εμφανιστούν θα είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ε, έλλειψη σαφήνειας ε, και για οποιαδήποτε εμπόδια παρουσιαστούν στη δουλειά των ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Φράγα. Καταρχήν μια γενική, ένα γενικό σχόλιο και μετά κάποια ειδικά, ειδικές παρατηρήσεις. Καταλαβαίνω την ε, βιασύνη. Μια και έχουμε αποφασίσει ότι την 1η του 2015 θα αρχίσει να εφαρμόζεται η ε, απαγόρευση απορρίψεων. Όμως, νομίζω ότι πάμε υπερβολικά γρήγορα εις βάρος της ίδιας της εφαρμογής του μέτρου. Η Κομισιόν αναγνωρίζει στην αιτιολογική έκθεση τη σχέση όλων αυτών με τα τεχνικά μέτρα και με την ανάγκη αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων. Εξηγεί η Κομισιόν την ανάγκη της μείωσης των απορρίψεων ε, διαμέσου της υιοθέτησης και της χρήσης ε, νέων ε, αλληλευτικών εργαλείων. Αυτό έκανε και η Νορβηγία. γιατί να μην τα κάνουμε όλα αυτά παράλληλα. Έχουμε μια καινούρια πρόταση, χωρίς όμως να ξέρουμε τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν για τα τεχνικά μέτρα. Όταν είδαμε τις τελευταίες αναθεωρήσεις του 850, τις νέες παρατάσεις δηλαδή, είχαμε πει ότι θα τροποποιήσουμε τον 850. Και είχαμε πει ότι οι επόμενες αναθεωρήσεις θα πρέπει να είναι συνολικές. Τώρα, ε, το impact assessment, τα impact assessment, ε, τις μελέτες ε, επιπτώσεων. Όταν είδαμε τις αντίστοιχες μελέτες για την κοινή αλληλευτική πολιτική, συζητούσαμε μια μεθοδολογία για τη μείωση των απορρίψεων στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Και από εκεί περάσαμε όμως σε μια απαγόρευση με συγκεκριμένες συνέπειες έγινε μελέτη συνεπειών για, το, για την απαγόρευση απορρίψεων. Διότι άλλο αυτό που τελικά αποφασίστηκε και άλλο το πώς είχαμε ξεκινήσει και με ποιες μελέτες επιπτώσεων είχαμε ξεκινήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτές οι αρχικές μελέτες επιπτώσεων χρησιμεύουν για να αναλύσουμε την τελική πρόταση. Πέστε μου, έχω δίκιο, φαντάζομαι να μου πείτε πως όχι, αλλά... Περνάμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα σημεία της πρότασης. Έχουμε και το χρονοδιάγραμμα βέβαια, αλλά το αφήνω για αργότερα. Μου, λέτε, μου λένε, δεν πρόκειται ε, μέχρι τον Απρίλιο να συνεδριάσει το Σύμβουλο Υπουργών Αλίας. Οπότε δεν πρόκειται να ληφθεί καμία απόφαση κατά διάρκεια αυτής της θητείας. Κανένα πρόβλημα. Το έχω συγχαθεί λιγάκι το θέμα αυτό. Στον 850, άρθρο 15.3 λέτε ότι οι καπετάνοι των αλλιευτικών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ε, πριν το ταξίδι ε, την πρόβλεψη των αλλιευμάτων. Και τι θα γίνει αν κάνει λάθος ένας καπετάνιος. Και τι χρησιμεύει αυτό το άρθρο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δεύτερο θέμα. Ε, η εξαποστάσεως ηλεκτρονική παρακολούθηση. Πολύ ωραία, ωραίο το άρθρο αυτό. αλλά πώς, σε ποιον και πού εφαρμόζεται. Ωραία όλα αυτά θεωρητικά, αλλά δεν δίνεται καμία πρακτική λεπτομέρεια για το πώς θα εφαρμοστεί, πού θα εφαρμοστεί και σε ποιον θα εφαρμοστεί. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δοθεί μια διευκρίνηση γι' αυτό. Μετά. Ε, άρθρο για την αποθήκευση στο πλοίο. Τι θέλετε να μας πείτε δηλαδή, ότι στη Μεσόγειο ένα πλοίο 12,5 μέτρα μήκος θα πρέπει να έχει διάφορα εργαλεία ε, και για κάθε είδος κάτω από το ελάχιστο μέγεθος να έχει ένα διαφορετικό ε, ε, κουτί όπου θα τα αποθηκεύει, πραγματικά αυτό είναι σαν να μας κάνετε πλάκα. Ωραίο χωρατό. Και μάλιστα τα πελαγικά είδη να είναι, ε, ε, τα βαθύβια είδη να είναι και χωριστά. Και μάλιστα να έχουν και ένα ε, πρόγραμμα ε, και αποθήκευσης απολύτως προσδιορισμένο και με λεπτομέρειες. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ αστεία. Δύνατο αυτό να γίνει στη Μεσόγειο. παραβάσεις και οι ποινές. Ωραία, σοβαρές οι παραβάσεις, αλλά ε, τι γίνεται με, τους, ε, το point system, ε, θα μείνουν οι ίδια, θα μείνουν οι ίδιοι πόντοι. Θα είναι διαφορετικοί Το 404 δεν τον αλλάζετε. Θα μου δώσετε μια εξήγηση για να κατάλαβω πώς θα λειτουργεί το point system. Θα αλλάξει κάτι στο 404. Ε, ελάχιστα μεγέθη μεγέθη αναφοράς. Δεν ξέρω γιατί αλλάζουν το όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει Στη Μεσόγειο βλέπω ότι δεν αλλάζει, δεν αλλάζουν τα μεγέθη, μόνο αλλάζει το όνομα. Ε, πάντως σε σχέση με το 850 κάποια αλλάζουν. Ε, ορισμένα μάλιστα ε, ήδη εξαφανίζονται. Και τι σχέση θα έχει αυτό με τα μεγέθη εμπορίας. Δεύτερον, ή τελευταίο, τι άλλο να σας πω. Α, εδώ βάζω τελεία. Πολλά προβλήματα εφαρμογής αυτής της πρότασης. Πού οφείλονται όλα αυτά, στη διασύνη μας. Στο Κορεπέρ ε, αλλά και στα περιφερειακά συμβούλια γίνεται πολλή δουλειά και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλή δουλειά, ιδιαίτερα στην Κορεπέρ, γιατί, για να καθορίσουμε καλύτερα τα πράγματα. Γιατί ε, και ο κλάδος και ο τομέας θα επιβαρυθούν πολύ. Και μου ξέχασα και κάτι άλλο. Κάτι άλλο η υποχρέωση της ατομικής αδειοδότησης των ε, εκφορτώσεων. Θα εφαρμοστεί τελικά σε όλα τα πλοία, σε όλα τα σκάφη. Τι νόημα έχει αυτό, δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα όριο μήκους για να μην αυξήσουμε τα βάρη ε, των ε, διοικητικών αρχών. Γιατί οι διοικητικές αρχές θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να διαχειριστούν τόσα καινούρια πράγματα επιπρόσθετα των όσων είχαν ήδη λόγω του κανονισμού ελέγχου. Τι είναι αυτά, αυτά είναι υποχρεώσεις που χρειάζονται ή δεν έχουν πολύ νόημα. Αυτές είναι δικές μου αμφιβολίες. Ας, τα, σκεφτούμε. Εγώ είμαι καλοπροαίρετη, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα θα έπρεπε να το είχαμε συνδέσει με τις τροποποιήσεις στα τεχνικά μέτρα. Αλλά αυτή τη στιγμή πάσχει από πολλές ασθένειες. Και όπως είπαν και πολλα κρατημέλη ε, μπορεί να οδηγήσουμε τον κόσμο τελικά να συνεχίσει τις απορρίψεις. Ε, Ζητώ συγγνώμη που πήρα τόσο χρόνο, αλλά ξέρετε, το, το έχω μέσα μου, στο αίμα μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευχή που εκφράσατε να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα με νυφαλιότητα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει έτσι όπως το είπατε, τουλάχιστον από πλευρά μου. Η Κομισιόν μας λέει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι δεδομένο. Αν σας κατάλαβα καλά, εκπρόσωπα της Επιτροπής. Αλλά το χρονοδιάγραμμα είναι βαθμιαίο. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρξουν πτυχές που πρέπει να διεκπαιρεώσουμε ταχύτατα, προφανώς, κυρίως τα απελαγικά είδη, γιατί έχουμε προθεσμία μέχρι την 1η Πρώτου 15. Κατά τα άλλα όμως έχουμε χρόνο να εκπονήσουμε με πιο προσεκτικό τρόπο τις ε, υποχρεώσεις. Γιατί οι υποχρεώσεις ε, θέτουν πολλά τεχνικά ερωτήματα και οικονομικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάποια προσωρινά πράγματα γρήγορα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ε, θα κρατήσουν και αυτά τα οποία θα είναι μακρόπνο θα πρέπει να τα δούμε με νυφαλιότητα. Για αυτό το χρονοδιάγραμμα υπάρχει λοιπόν αυτή η πρώτη αντίφαση. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην αιτιολογική σκέψη και στην πρόταση του τροποποιημένου κανονισμού. Γιατί στην αιτιολογική σκέψη του α, κανονισμού, στην σελίδα 2, σημείο 4, λέτε «Εν, εν αναμονη του νέου πλαισίου θα πρέπει προσωρινά να υιοθετήσουμε ε, νομοθετικά μέτρα, ε, ακυρώνοντας τα νομοθετικά εμπόδια που μπορεί να θέσουν ένα αμφιβόλο αυτή την υποχρέωση, δηλαδή εκφόρτωση εννοεί, υποχρέωση εκφόρτωσης. Μιλάμε για μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 15, λοιπόν. Σε όλο τον κανονισμό, εν συνεχεία, και όχι πια στην αιτιολογική σκέψη, σε όλο τον υπόλοιπο κανονισμό υπάρχουν αναφορές στο άρθρο 15, ήδη στο μεταβατικό κανονισμό, και για τα πελαγικά είδη και για όλα τα υπόλοιπα αλλιεύματα ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα. Επομένως, δεν μιλάμε για καμία βαθμία προσέγγιση. Ε, αυτό ισχύει για όλο τον κανονισμό. Δηλαδή εφαρμόζουμε το άρθρο 15 σε όλο τον κανονισμό με τις προθεσμίες που αναφέρονται στο βασικό κανονισμό. Αυτό είναι πρόβλημα. Θα πρέπει τα πράγματα να τα πούμε ξεκάθαρα γιατί έχουμε να κάνουμε ένα κανονισμό ο οποίος αφορά και τα κατεπήγοντα και την υποχρέωση ε, εκφόρτωσης για τα περιλογικά είδη από τη μία ή μήπω έχουμε να κάνουμε για ένα γενικό κανονισμό που αφορά όλα τα είδη και επομένως είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό ως παρατηρήσει για την προθεσμία, για τις προθεσμίες. Τώρα, δύο-τρία σχόλια εντάχει ε, υποτύπων ερωτήσεων. Καταρχάς, συμφωνώ με την Κάρμεν Φράγκα για τις προβλέψεις ε, αλλιευμάτων. Ε, τι έπαθαν εδώ οι συντάκτες, ε, τους ήρθε παλήρια στα μούτρα. Επίσης, δεν σκέφτεστε καθόλου διαφορετικές ε, δυνατότητες, εναλλακτικέ δυνατότητες, πέρα από την βίντεο επιτήρηση. Γιατί αυτή είναι μία τροχοπέδη στην ελευθερία εργασίας μέσα σε καλές συνθήκες. Ας το σκεφτούμε, μήπως υπάρχουν και άλλες τεχνικές λύσεις, όχι μόνο βίντεο παρακολούθηση. Δηλαδή, επειδή σκεφτόμαστε πιεσμένοι χρονικά, ε, σκεφτόμαστε μόνο ένα μέτρο τεχνολογικό, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα τεχνολογικά μέτρα. Η επιλεξιμότητα, η επιλεκτικότητα μάλλον. Εγώ δεν ξέρω αν έχω καταλάβει καλά την, την υπόθεση της εκφόρτωσης απορρίψεων. Το θέμα δεν είναι να εκφορτώνουμε, το θέμα είναι να πιάνουμε ό,τι έχει εμπορική αξία. Αυτό είναι το βασικό. Ο βασικός στόχος για μένα είναι η επιλεκτικότητα. Εδώ μιλούσαμε για το άρθρο ε, του 850 θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άρθρο που διευκολύνει την επιλεκτικότητα. Συμφωνώ ότι θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες τεχνικές δυσκολίες σε αυτόν τον κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα, ε, τα κατεπήγοντα, πρώτη Πρώτου 2015 για την εκφόρτωση των ε, πελαγικών ειδών και πιο νυφάλια, πιο ήρεμα για όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πολύ με τους προλαλήσαντες ότι το πιο σημαντικό πράγμα κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης απορρίψεων είναι να εμποδίζουμε τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα και γι' αυτό ελπίζω η Task Force μας να σημειώσει πρόοδο κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Το θέμα επίγει. Πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα όσο βρισκόμαστε εδώ, οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις αυτές με το Συμβούλιο. Στο σχέδιο διαχείρισης λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις για να αποφευθούν τα παρεπίπτωτα λιεύματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εξίσου σημαντικό θα έλεγα είναι το θέμα του ελέγχου. Χωρίς έλεγχο Μπορεί να λέμε πολλά ωραία λόγια στα νομοθετήματα, εάν όμως κανείς δεν ελέγχει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τότε τα πράγματα θα συνεχιστούν ως έχουν. Οι διατάξεις ελέγχου λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τρίτον, ε, θα ήθελα επίσης να αναφέρω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι Όλοι εδώ μιλούν μόνο για τα πελαγικά είδη για το 2015. Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Μιλάμε για το σύνολο της Βαλτικής θάλασσας. Μιλάμε δηλαδή για Σολομό, μιλάμε για Γάδο στη Βαλτική. Ξέρω ότι ο Περιφερειακός Φορέας που το συζητάει αυτό αναφέρεται και στην ε, θαλάσσια απέστροφα, την ε, Σαρδελόρεγκα τη ρέγγα και το γάδο. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τα πελαγικά είδη. Έχω κάποιες δύσκολες ερωτήσεις. Μου φαίνεται ότι στις συζητήσεις για τη Βαλτική κάποια κράτη θέλουν να συμπεριληφθούν επιπλέον είδη, άλλα όχι. Δεν ξέρω πώς αυτό σχετίζεται με την πρόταση της Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 στον βασικό κανονισμό, τα κράτη-μέλη μπορούν να προτείνουν είδη τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται από την υποχρέωση εκφόρτωσης σε πέρα από τα είδη που ήδη αναφέρονται. Αλλά εάν κάποιο κράτος θέλει να συμπεριλάβει ένα είδος και κάποιο άλλο όχι, θα επιτρέπετε κάτι τέτοιο, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην περίπτωση αυτή. Επίσης, ε, θα είναι δυνατόν για τα κράτη-μέλη να αποκλείσουν κάποια είδη εξοπλισμού από την υποχρεωσία εκφόρτωσης. Αυτές είναι οι γενικές ερωτήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες του τεχνικού κανονισμού είναι φυσικά πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζω ότι θα πρέπει να εργαστούμε γρήγορα πάνω στο θέμα αυτό, διότι η υποχρέωση εκφόρτωσης στη Βαλτική θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, για την παρέμβασή σας. Ε, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Είναι πολύ αντικειμενικά τα θέματα. Βασίζονται στην ε, κοινή αλλιευτική πολιτική που υιοθετήσαμε πριν κάποιους μήνες. Απογοητευτικό. Είναι ότι δεν υπάρχει κίνητρο παρά μόνο για τους αλληλείς ε, να μην αλλιεύουν τα παρεμπιπτόντα αλλιεύματα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Σήμερα ασχολούμαστε με τα τεχνικά μέτρα κανονισμού την ε, τροποποίηση των σχετικών ε, του σχετικού κανονισμού. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν. Δεδομένου ότι προτείνεται να εισαχθεί απαγόρευση απορρίψεων για τα πελαγικά είδη από την 1η Ιανουαρίου του χρόνου. Είναι δυνατόν να γίνει διαφοροποίηση ανάμεσα στα πελαγικά και τα άλλα είδη. Και αν ασχοληθούμε πρώτα με τα πελαγικά είδη, αυτό θα είναι πλεονέκτημα. Και επίσης, αν δεν γίνεται αυτό, ε, ποια είναι η εναλλακτική λύση που προτείνει η Κομισιόν, το σχέδιο Β. Ο κύριος Κρίστενσεν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε υιοθετήσει τώρα μία ε, αλλιευτική πολιτική με το βλέμμα στο μέλλον, με περισσότερη βιωσιμότητα. Θέλουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο των αλλιευμάτων στις θάλασσες. Τους τελευταίους μήνες έχω συνομιλήσει με αλλιείς στη Δανία και Όταν ακούν ότι θα ελέγχουμε περισσότερο τα μέτρα, ανησυχούν οι αλήσει στη Δανία. Διότι έχουν πολλούς κανόνες ελέγχου με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφωθούν. Αυτή λοιπόν η αλλιευτική πολιτική, εάν απαιτεί περαιτέρω μέτρα ελέγχου, όπου λόγω της εκφόρτωσης όλων των ψαριών ε, θα πρέπει να μειώνεται το άχθος ε, ελέγχου, πιστεύω ότι θα πετύχει αυτή η μεταρρύθμιση. Στους ελείς και στις ε, περιφέρειες έχουμε υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε τη θέση τους με τη διαδικασία της περιφερειοποίησης, διότι διαφέρει η αλληλεία στις διάφορες θάλασσες της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν, η περιφερειοποίηση αυτή πώς θα πραγματοποιηθεί. Δεν πρέπει να ακούσουμε τους ενδιαφερομένους στις διάφορες περιφέρειες, ώστε να ληφθεί υπόψη η γνώμη τους κατά διαμόρφωση των κανόνων. Εννοείται ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να είναι σαφείς οι κανόνες. Να μην υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία και θα υπάρξουν εάν δεν το κάνουμε αυτό. Στον ένα κανονισμό δηλαδή θα επιτρέπεται η απόρριψη κάποιων ειδών, σε άλλον κανονισμό θα απαγορεύεται η απόρριψη και αυτό δεν θα λειτουργήσει στη πράξη. Πρέπει οι κανόνες να είναι σαφείς. Πιστεύω όμως ότι είναι σαφές. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν με καλό τρόπο όλα αυτά, ώστε να νιώθουν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικής ώστε να έχουμε μακροπρόθεσμα μία βιώσιμη πολιτική, την οποία να υποστηρίζουν όλοι. Ευχαριστώ. Bien, muchas gracias. Ninguna otra intervención. Damos la palabra a la Comisión. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Δύο preguntas y cuestiones. Να απαντήσει αυτό το μακρύ και εκτενή κατάλογο με ερωτήσεις. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις ε, για να απαντήσω καλύτερα, όπου μπορώ. Να ξεκινήσω όμως από το τελευταίο σχόλιο που έγινε για την περιφερειοποίηση. Δεν το έκανε μόνο ο τελευταίος ομιλητής και κάποιοι άλλοι πριν. Θα θυμάστε, όπως είπε η κυρία Αρντεβίν, ότι στη νέα κοινή αλληλευτική πολύ ε, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να ενεργοποιήσουμε την περιφερειοποίηση. Ε, τι γίνεται ανάμεσα στην ε, σημερινή χρονική στιγμή και στην ε, μελλοντική στιγμή. Ελπίζουμε να υπάρχει δυνατότητα πιο επιλεκτικής αλίας. Το κίνητρο της επιλεκτικής αλίας μπορεί να ρυθμιστεί στο πλαίσιο των σχεδίων ε, απορρίψεων. Και αυτό μπορεί να γίνει με την εμπλοκή των αλλιέων, των συμβουλευτικών οργανώσεων και των ορμάδων, ούτως ώστε για κάθε μορφή αλίας, για κάθε αλίευμα να έχουμε την κατάλληλη απάντηση. Εσείς επειδή εμπλακήκατε σε διαπραγματεύσεις για τεχνικά μέτρα, εδώ στις Βρυξέλλες ξέρετε ότι τεχνικά είναι δύσκολο και ότι χρειάζεται πολύ χρόνο. Χρόνο που δεν έχουμε. Γι' αυτό ακριβώς η προσέγγιση που παρουσιάζουμε εδώ, και εδώ μπαίνω σε ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε, είναι να εξασφαλίσουμε ότι προς το παρόν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Η κυρία Τομάου μίλησε για τους κανόνες που θα ισχύσουν για την εκφόρτωση και τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι κανόνες. Θα είναι απλή διόρθωση ανάμεσα στο σήμερα και στην τελευταία φάση της θέσης ισχύς της υποχρέωσης ε, ε καθαρίσεων, ε, εκφορτώσεων, ε, ο 850, όπως τροποποιείται από μας σήμερα, θα είναι η βάση για να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης στην πρώτη φάση. Και ενώ θα προχωρούμε προς τη δεύτερη και τρίτη φάση, θα έχουμε ελπίζουμε, μία συμφωνία που θα επιτρέπει ε, μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης με περιφερειοποίηση. Τα νέα, το νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων. Όταν θα έχουμε το νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων, που θα έχει διαπραγματε... διαπραγμάτευση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τότε αυτό πριτανεύει σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε για το 16, 17, 18, 19. Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα πλαίσιο, κολλάνε. Δεν θέλουμε να συμβεί το εξή, κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και μπορεί να ξανασυμβεί, όπου οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τα νέα τεχνικά μέτρα κρατάνε πάρα πολύ. Και βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, ας πούμε, του 2015, όπου χρειαζόμαστε τελευταία στιγμή μια ακόμα πρόταση μέσα σε απελπισία, ούτω ώστε να μην βρεθούμε σε δυσκολία μέχρι την πρώτη κυρία δυο επιπεδα όπω ειπε η κυρια φραγκα Οι γρήγορε λύσει και οι μακρόπνοε ε, λύσει. Αλλά οι γρήγορε λύσει ε, ισχύουν μόνο και μόνο για να άρουν τις φοβερέ αντιφάσει στην ε, νομοθεσία. Δεν προδικάζουν αυτό που μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη και οι αλληλείς περιφερειακά μέσω των σχεδίων απορρίψεων. Και τη δουλειά θα κάνετε εσείς το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο για την υιοθέτηση των νέων τεχνικών μέτρων. Ο κίνδυνος, ο Τομάς, είναι να έχουμε παράλληλες διαπραγματεύσεις τελικά για τα νέα, το νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων του χρόνου και την προσπάθεια ευθυγράμμιση ε, των κανόνων. Α πούμε ότι είμαστε 1η Ιουλίου του 2015. Εσεί διαπραγματευόστε με το Συμβούλιο για τα νέα τεχνικά μέτρα. Θα πρέπει να διαπραγματευτείτε και, μια και δεν θα υπάρχει αρκετό χρόνο για να εξασφαλίσετε την υιοθέτηση των νέων κανόνων μέχρι 1η του 2016, πρέπει να διαπραγματευτείτε ένα άλλο νομοθέτημα παρόμοιο με αυτό, παράλληλα. Κάποια στιγμή δηλαδή μπορεί να έχετε να κάνετε δύο πράγματα και να πιεστείτε ακόμα περισσότερο. Και αυτό μπορεί να δυσκολεύσει πολύ την κατάσταση. Γι' αυτό που είπε η κυρία Φράγκα για τη μελέτη αντικτύπου. Αυτή η πρόταση που κάνουμε δεν βασίζεται σε μια νέα μελέτη αντικτύπου. Σωστά το είπε η κυρία Φράγκα. Γιατί δεν την κάναμε όμως. Ξέρετε, λόγω χρονικής πίεσης. Αλλά όχι μόνο. Γιατί και αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτά που εσείς αποφασίσατε με το Συμβούλιο τα μεταφράζουμε σε ένα κείμενο. Δεν είναι μια νέα πολιτική, είναι μια τεχνική ευθυγράμμιση των κανόνων, ούτω ώστε να άρουμε τις ασυνέπειες. Γιατί αλλιώς θα έχουμε μια νομοθεσία που θα λέει θα πρέπει να εκφορτώνεται και μια άλλη που θα λέει θα πρέπει να απορρίπτεται. Γι' αυτό η κανονική μελέτη αντικτύπου που κάνουμε όταν κάνουμε μια νέα πρόταση που αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο εν το βάθη, επί της ουσίας, δεν έχει γίνει. Η κυρία Φράγκα επίσης μίλησε και για άλλα πράγματα, όπου το κείμενο μπορεί να βελτιωθεί, σωστό. Περιμένουμε τα σχόλια και τη σοφία της Επιτροπής σας. Ούτως ώστε αυτή η αυτό ο εξορθολογισμό του συστήματος να γίνει πραγματικότητα. Αυτή η ευθυγράμμιση να γίνει πολύ καλύτερη. Η κυρία Φράγκα αναφέρεται στον κανόνα που αφορά τους καπετάνιου καπετάνιους, ότι θα πρέπει να προβλέψουν τις, την αλίευση που θα κάνουν, τα αλίευματα. Μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό το σημείο. Επίσης, για τις, τα πολλαπλά είδη αλιευμάτων στη Μεσόγειο θα πρέπει να έχουμε διαφορετικό κουτί όπου θα στηβάζουμε κάθε είδος. Ίσως όχι. Επίσης, πώς θα αποφύγουμε τη γραφειοκρατία στις εθνικές διοικήσεις. Και εδώ μιλάω για τις μεμονωμένες αδειοδοτήσεις. Καλώς όλοι αυτά τα σχόλια. Πραγματικά βελτιώνουν το κείμενο. Θα το βελτιώσουν τελικά. για τις κάμερες. Αυτό που λέει το κείμενο είναι ότι έχουμε κάποιους ε, τρόπους ε, ελέγχου στον κανονισμό ελέγχων, ε, επιθεωρήσεις πάνω στο σκάφος και το συμπληρώνει αυτές τις διατάξεις. Μιλάει για CCTV. Δεν είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου άρθρο 15 και υποχρέωση εκφόρτωσης. Δεν είναι μόνο το κλειστό κυκλώμα τηλεόραση στο CCTV. Όχι. Ξέρουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει, σε ορισμένα κράτη-μέλη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κλειστά κυκλώμα τηλεόραση. Για κάποιε μορφέ αλληλεία. Γιατί υπάρχει συμφωνία για τη χρήση του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά. Είναι κάτι που προστίθεται σε μια σειρά άλλων μέτρων που διαθέτουμε ήδη. Ελέγχου. για την επιλεκτικότητα. Το, το σχολίασα. Πώς τη διευκολύνουμε την επιλεκτικότητα. Ε, συνεργαζόμαστε με, τα, με τις περιφερειακές οργανώσεις με τις εμβουλευτικές οργανώσεις και ελπίζουμε να συμβουλεύσουν τα κράτη-μέλη για καλά σχέδια απορρίψεων. Τα καλά σχέδια ποια είναι. Αυτά, αυτά που λαμβάνουν υπόψη είναι αυτά που είπατε πολλοί από εσά. Ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τελικά ασχολούμαστε με τα αλλιεύματα. Επομένως η αποφυγή και η επιλεκτικότητα είναι πολύ σημαντικά θέματα. Να αποφεύγουμε να πιάνουμε είδη που δεν μας ενδιαφέρουν. Η κυρία Λεβίν επίσης έκανε μια αναφορά στη Βαλτική, όπου κάποιες χώρες μπορεί να θέλουν να συμπεριλάβουν και άλλα είδη. Ο τρόπος για να βάλουμε κανόνες άχρηστούν είναι τα σχέδια απορρίψεων. Γιατί προς το παρόν Δυστυχώ τα πολιετή σχέδια είναι μπλοκαρισμένα. Ελπίζω για, όχι για πάντα, όχι για πολύ, αλλά δεν υπάρχει. Η κυρία Λεβίν ρώτησε επίση αν μπορούν να αποκλείσουν τα δρανή εργαλεία τα κράτη-μέλη. Όχι. Το κύριος Γκάλαγκερ ρώτησα κάποια πράγματα, ελπίζω να σας απάντησα. Μας ρωτήσατε αν τελικά, στο τέλος του χρόνου, δεν υιοθετηθούν όλα αυτά. Υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Η μόνη που μπορώ να σκεφτώ τώρα είναι ότι θα πρέπει να συζητήσουμε με τις εθνικές αρχές και να εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές, διευκρινιστικές μη δεσμευτικές, που θα εξηγούν τους εφαρμοστέους κανόνες. Ένα είδος, ας πούμε, χειριδίου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ψαράδες, από τους επιθεωρητές και από τις εθνικές αρχές και να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Είναι η μόνη εναλλακτική λύση που βλέπω, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε νομοθεσία αν δεν θέλουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεν είναι το τέλειο, αλλά τουλάχιστον θα υπάρξει μια διευκρίνηση στους εφαρμοστέους κανόνες. Ελπίζω να σε απάντησα σε όλα. Και να προσθέσω και ένα τελευταίο. Θα κυκλοφορήσουμε ένα πίνακα αντιστοιχήσεις που μπορεί να βοηθήσει τη δουλειά σας, όπου θα περιγράφει λεπτομερώς για κάθε μία από τις διατάξεις που υπάρχουν, σε τι αναφέρονται, τι αλλαγές επιφέρουν κτλ. Και ελπίζω να σας βοηθήσει. Πρόεδρος, είναι δύσκολο να συνδυάσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, την πολυπλοκότητα. Δεύτερον, την απαραίτητη ταχύτητα. Επιπλέον, διαφωνώ με κάποια πράγματα που είπε η Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν υπερβαίνει την απαραίτητη τεχνική ευθυγράμμιση ε, ζήτησε, λέει ότι απλώς προσπαθεί να διορθώσει αλογικές ασυνέπειες. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα θα ήταν εύκολο, αλλά υπερβαίνει αυτά που είπε η Κομισιόν. Είναι αλήθεια ότι έχουμε περιορισμό, αρχικό περιορισμό χρόνου που είναι η 1 πρώτη του 2015 και το γεγονό ότι δεν περιοριζόμαστε τα πελαγικά είδη ε, όλα αυτά περιπλέγουν την κατάσταση, αλλά είναι αλήθεια πως, ε, όπως είπε η Κομισιόν, ε, δεν επιθυμεί να ε, αντιμετωπίσει το θέμα των τεχνικών μέτρων συνολικά, γιατί πιστεύει ότι το 2016 δεν θα είναι έτοιμα και θέλει όλα αυτά να τα δει σταδιακά. Δεν το Δεν συμφωνώ με αυτό καθίστε να δουλέψετε, σηκώστε τα μανίκια, να τα σηκώσουμε κι εμείς, έτσι ώστε να τα καταφέρουμε έστω και με παράλληλε διαπραγματεύσει αλλού. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι την 1η 2015. Θα πρέπει από τώρα να στρωθούμε στη δουλειά. Τούτου λεχθέντος πραγματικά ειλικρινά δεν γνωρίζω δεν, ε, δεν είμαι σίγουρος, αλλά υποπτεύομαι πως η Κομισιόν έχει επωφεληθεί αυτής της διαδικασίας για να περάσει και άλλα μέτρα. Δεν είμαι σίγουρος για το μέχρι πού θα μπορούσαμε να φτάσουμε όμως. Μέχρι τον Απρίλιο, πριν τις εκλογές. Μετά θα έχουμε καινούργια επιτροπή αλήθεια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί. Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνοδεύσει αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Οπότε δεν ξέρω τι θα προκύψει από το καινούριο κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να πάρουμε μια απόφαση, γιατί ε, υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες από ό,τι ε, φαινόντουσαν σε πρώτη προσέγγιση. Η εντύπωσή μου και η εντύπωσή μας είναι ότι ε, δεν θα το καθαρίσουμε εύκολα αυτό το θέμα δίνοντας λευκή επιταγή στην Κομισιόν. Οπότε θα προτείνω και το προτείνω ήδη ε, ένα χρονοδιάγραμμα συνεδριά συνεργασία μαζί με τους κοιόδης ενδεχομένω για να προγραμματίσουμε το πώς θα χειριστούμε αυτή την έκθεση. Την έχω αναλάβει εγώ μόνο ως πρόεδρος και όχι ως εκπρόσωπος κάποιας πολιτικής ομάδας. Το σημαντικό είναι να το δούμε όλοι μαζί. Θέλει κανείς να πει κάτι. Κυρία Τομά. Oui, Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήθελα να ξαναπάρω το λόγο, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα ήρεμο και επικοδομητικό διάλογο, θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά και τίμια. Στο θέμα για την βίντεο παρακολούθηση, κομισιόν μου απαντάτε ότι δεν είναι υποχρέωση κάτι τέτοιο και ότι θα ισχύσει ανάλογα με τη χώρα. Διαβάζω το 25β του α για την ε, εξαποστάσεως βιντεοπαρακολούθηση. Ένα λευτικό σκάφο που δυνάμει τη νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μια απόφαση που υιοθετήθηκε από ένα κράτο μέλος, δεν είναι και ένωση και κράτος μέλος, είναι ή ένωση ή κράτος μέλος. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ε, εξ αποστάσεως ηλεκτρονική παρακολούθηση για να ελέγξουν την υποχρέωση εκφορτώσεων κτλ. Θα πρέπει να έχουν τα, το απαραίτητο εξοπλισμό, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός. Α. Ε, διάταξη ε, που θα πρέπει να εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές, όλες οι εικόνες και οι αληφτικές δραστηριότητε φυλάσσονται μονίμως. Δεν είναι μια άδεια που δίνουν τα κάτι μελη μερικά τη δίνουν, μερικά όχι. Όχι, μέχρι στιγμή είναι το μόνο μέσο ελέγχου το οποίο προβλέπει η τροποποίηση του 850. Και θα γενικευθεί. Ή μάλλον δεν καταλαβαίνω καλά, ή αν, δεν καταλαβαίνω, ή αν εγώ δεν καταλαβαίνω καλά, έχετε λάθος διατύπωση. Πρέπει να την αλλάξετε. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να μας πουλήσετε κάτι ψεύτικο. Ας μην κάνω παρομοίωσεις εδώ και μεταφορές. Έτσι. Πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά και τίμια. Ευχαριστώ κύριε Τωμά. Ο κύριος Γκάλαγκερ. Πρόεδρε, όλοι θέλουμε να εφαρμοστεί η απαγόρευση απορρίψεων από την 1η Ιανουαρίου του 2015, αλλά η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι η πελαγική αλίεν είναι πολύ πιο καθαρή από ότι πολλά είδη πελαγικής, όταν μιλάμε για διάφορα είδη ρέγκας και σκουπριού. Υπάρχει όμως κάποιο όφελος, εάν επικεντρωθούμε σε αυτό από 1η Ιανουαρίου του 2015 ή είναι καλύτερα να καθυστερήσουμε και να ασχοληθούμε με όλα τα είδη παράλληλα. Εκτιμώ αυτό που είπε η Κομισιόν, αλλά το σχέδιο Β είναι μόνο κατευθυντήρες γραμμές, ε, δεν είναι υποχρεωτικές. Εάν υιοθετηθούν από 1η Ιανουαρίου οι κατευθυντήρες γραμμές, εάν ο κανονισμός υιοθετηθεί 1η Ιανουαρίου, για παράδειγμα, από όλα τα θεσμικά όργανα, τι θα γίνει. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε την 1η Ιανουαρίου 2015 ε, την απογόρευση για την πελαγική αλία. Άλλες παρεμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρητικά είναι δυνατό να εστιαστούμε στα πελαγικά είδη, αλλά έχουμε και τη βαλτική. Αν σαλαμοποιήσουμε τα μέτρα, θα δούμε τα βενθοπελαγικά, αλλά ε, θα πούμε στο, στο αδιέξοδο ότι θα πρέπει να προβλέψουμε τι θα γίνει για τα βενθοπελαγικά αλλού σε άλλες διαπραγματεύσεις. Ίσως θα διευκόλυνε λίγο, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε πολλές πολλά στοιχεία που περιπλέκουν την κατάσταση. Αν μπορώ να συνεχίσω στα γαλλικά, ε, κυρία Τωμά, δύο λόγια. Δεν προσπαθώ να σας κοιμήσω με τεχνικές λεπτομέρειες. Ίσως δεν έχει γραφτεί καλά, αλλά ο στόχος του κειμένου είναι να προσθέσουμε κάτι το οποίο λείπει στον σημερινό κανονισμό ελέγχου τα μέτρα ελέγχου που υπάρχουν θα συνεχίσουν να υφίστανται. Ε, η παρακολούθηση ε, από το σκάφος ε, θα μπορέσει να συνεχίσει να εφαρμόζεται, να χρησιμοποιείται. Δεν το βάλαμε, διότι θέλουμε να προσθέσουμε με αυτό το κείμενο. Δεν αναφερόμαστε πράγματα που υπάρχουν ήδη. Με το κείμενο το οποίο σας υποβάλλουμε θέλουμε να προσθέσουμε. Προσθέτουμε τεχνικές προδιαγραφές ή θέλαμε να προσθέσουμε τεχνικές προδιαγραφές που λείπουν αυτή τη στιγμή από τον νόμο. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο δηλαδή ένα κράτος μέλος, αποφασίσει ότι το καλύτερο μέσο να ελέγξουν την, ε, την απαγόρευση ε, απορρίψεων είναι οι κάμερες. Έτσι εμείς θέλαμε, αυτή, αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Όχι να καταστήσουμε μέσω αυτού του κειμένου υποχρεωτική τη χρήση καμερών. Επί των αλληλευτικών σκαφών. Είναι κάποιες τεχνικές προδιαγραφές μόνο, αυτές που προτείνουμε, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που η ευρωπαϊκή εθνική νομοθεσία απαιτήσει την χρήση καμερών. Ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή μας. αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, κλείνουμε αυτό το θέμα, περνάμε στο επόμενο θέμα της μεσίας διάταξης. Παρουσίαση από το θεματικό τμήμα Β του ενημερωτικού σημειώματο με θέμα η χρήση διατάξεων συγκέντρωση χθείων στην αλία τόνου. Το ενημερωτικό αυτό σημείωμα ανατέθηκε στην Scott Fishery Consultants. Έχετε το σημείωμα στα χέρια σας. Καλωσορίζουμε τον συντάκτη του σημειώματος, τον κύριο Jerry Scott και του δίνουμε το λόγο για να μας το παρουσιάσει. Έχετε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που μπορώ να σας ε, μιλήσω για τη χρήση των διατάξεων συγκέντρωσης χρήων ε, κατά την αλληλεία τόνου. Ελπίζω να λειτουργήσει η τεχνολογία. Στόχος λοιπόν της μελέτης αυτής ε, είναι να συνοψίσουμε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες όσον αφορά τη χρήση των διατάξεων αυτών ε, σε σχέση με την ικανότητα των ε, σκαφών να αλλιεύουν ψάρια. Βασίσαμε την ανάλυση αυτή στα δεδομένα που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης Αλληλείας. Εξετάσαμε τα δεδομένα αυτά και εξετάσαμε και άλλη βιβλιογραφία ε, και μιλήσαμε με εμπειρογνώμονες. Ε, εξετάσαμε τον βαθμό στον οποίο συνεχίζει να αυξάνεται η αλληλεία. Εξετάσαμε τις συνέπειες σε άλλα είδη και συντάξαμε και μια σειρά συστάσεων ε, που θα μπορέσετε να εξετάσετε. Πλωτές συσκευές ε, χρησιμοποιούνται εδώ και εκατοντάδες χρόνια για να βοηθήσουν τους αλληλείς ε, να αλλιεύουν ψάρια. Αλλά μόνο τα τελευταία 20 με 25 χρόνια η χρήση τροποποιημένων ε, πλωτών συσκευών έχουν χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσουν την ικανότητα των σκαφών να αλλιεύουν τόνο. Είδαμε μια μεγάλη σειρά καινοτομιών κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος και είδαμε αύξηση της ε, δυνατότητας ε, της αλίας με γρηγρή και κατόπιν είδαμε και ε, τον τρόπο αλίευσης τόνου με διατάξεις συγκέντρωσης ηχθείων. Υπάρχουν προσπάθειες να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες της αλληλέία με διατάξη για των και θα αναφερθώ σε αυτές σύντομα. Δύο ήδη υπάρχουν. Έχουμε τα πλωτά φαντς και έχουμε αυτά που είναι αγκιστρωμένα στο βυθό. Στόχο έχουν συνήθως να βοηθήσουν ε, τα, την ε, αλία μικρής κλίμακας ή την ημιοβιχαμνική. Ενώ ε, ε, οι αγκιστρωμένες χρησιμοποιούνται για την αλία βιομηχανικής κλίμακας. Γενικά χρησιμοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα. Εδώ βλέπετε μια γενική εικόνα επάνω της κατανομής ε, των σταθερών ε, ΦΑΤ. Υπάρχει μεγάλος ε, αριθμός στον Ινδικό ωκεανό αλλά και στη Μεσόγειο. Επίσης βλέπετε στη μέση κάποιες φωτογραφίες και ένα σχέδιο των ΦΑΤΣ και χρησιμοποιούνται και κάποιες ε, σημαδούρες ανείχνευσης ωκεανογράφων και έχουν υπάρξει κάποιες ε, αντιρρήσεις ε, σχετικά με τη χρήση τους. Και εδώ βλέπετε την κατανομή των πλωτών και την κατανομή τους. Οι δύο εικόνες κάτω δείχνουν ε, την βασική δομή. Αριστερά βλέπετε ότι υπάρχει μία ε, δομή που κρέμεται από μία πλωτή πλατφόρμα και είναι συνδεδεμένη μία σημαδούρα ηλεκτρονική εδώ που ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα. Δεξιά βλέπετε πώς φαίνεται από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόσφατα διάβαζα σε ένα blog για μια επιχείρηση στον Ειρηνικό όπου οι Αλείς συνάντησαν ε, μια νεκρή φάλαινα και κρέμασαν από τη φάλαινα κάποιον εξοπλισμό και έτσι την μετέτρεψαν σε φαντ. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν ε, πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία εμφανίζονται φυσικά στον ωκεανό ή που έχουν τοποθετηθεί από ανθρώπους. Εδώ βλέπετε άλλες εικόνες πιο πρόσφατων ΦΑΤ και κάποια έχουν στόχο να μετριάσουν το φαινόμενο του να μπλέκονται άλλα είδη στα δίκτυα. Συχνά, αν υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο να κρέμεται από το φαντ αυτό, ε, βλέπουμε συχνά ότι μπλέκονται στα δίκτυα είδη στα οποία δεν στοχεύουμε ιδιαίτερα καρχαρίες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια τεχνικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να μετριάσουν το πρόβλημα αυτό, αυτού του είδου, δηλαδή την θνησιμότητα, που γενικά δεν απαντάται στο είδο αυτό τη αλεία. Τα τρία είδη που ε, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εδώ είναι η παλαμίδα, ο κυθρινόπτερο και ο μεγαλόφθαλμος τόνος κάτω στο κέντρο. Από τα τρία αυτά είδη η παλαμίδα είναι αυτό που αναπτύσσεται πιο γρήγορα, ζει όμως λιγότερο. Συζητιέται το ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος, αλλά 18 κιλά ε, είναι το μέγιστο που υπολογίζεται συνήθως, ενώ στο αλίευμα ε, ζυγίζουν 3 με 5 κιλά. Ε, στα γρηγρή αυτό είναι το βάρος, εάν όμως αλλιεύουμε με φαντ, δηλαδή αν ε, ψάχνουμε για ε, ελεύθερα κοπάδια και συνήθως ε, έχουμε μεγαλύτερα ψάρια. Επίσης ο κυτρινόπτερος τόνος και ο μεγαλόφθαλμος πιάνονται και με παραγαδιάρικα όπου γενικά αλλιεύονται μεγαλύτερα ψάρια περίπου ενός μέτρου μήκους. Εδώ στην επάνω σειρά βλέπετε το μήκος των αλλιευμάτων που έχουν αλλιευθεί με φάτ στον Ειδικό Ωκεανό τα τελευταία χρόνια. Όπως βλέπετε και για τα τρία είδη, ε, συνήθως το μήκος είναι 50 εκατοστά, που στην περίπτωση της παλαμίδας ε, σημαίνει ότι πιάνουμε ενήλικα ψάρια, ενώ για τον κυτρινόπτερα και ε, τον μεγαλόφθερμο τόνο είναι μικρότερο από το μέγεθος των ενήλικων ψαριών, δηλαδή πιάνουμε μικρά ψάρια. Επίσης, βλέπετε εδώ ότι έχουμε στη μεσαία σειρά ότι έχουμε και ενήλικα ψάρια και ε, νεαρούς θαλασσούς οργανισμούς, ε, ενώ στον ε, μεγαλόφθαλμο βλέπετε ότι η αλία με φάντε έχει γίνει ο βασικός τρόπος αλίας τροπικών τόνων. Η αλία με φάντα έχει αυξήσει τη δυνατότητα των σκαφών να αλλιεύουν ψάρια. Ε, έχουμε αυτό που ονομάζουμε μυστική αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας, ε, δηλαδή ε, βελτίωση της ικανότητας αλίας με τεχνολογικές βελτιώσεις. Οι περισσότεροι αλληλείς πάντα θέλουν να πιάσουν περισσότερα ψάρια και Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αύξηση αλληλευτικής προσπάθειας σε πολλά είδη αλληλείας και στην ε, αλληλεία με παραγάδια για παράδειγμα. Στην περίπτωση των FAD, το βασικό χαρακτηριστικό μάλλον ε, είναι η τεχνολογική βελτίωσή τους ηλεκτρονική, βελτίωση στις ηλεκτρονικές σημαδούρες που συνδέονται με αυτά και η δυνατότητα ανείχνευσης ε, του τι κινείται κάτω από την ε, διάταξη συγκέντρωσης ηχθείως, καθώς και η χρήση βοηθητικών ε, σκαφών. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία σε αυτό το τεχνολογικό παιχνίδι. Οι πλωτήρες ανείχνευσης αποτελούν ε, την πιο σημαντική τεχνολογική ε, βελτίωση που έχει ε, πραγματοποιηθεί τα τελευταία 20 με 30 χρόνια για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αλίας τόνου. Ξέρουμε ότι αυτές οι καινοτομίες και σε επίπεδο σκάφους και σε επίπεδο στόλου ε, αναλαμβάνονται πολύ γρήγορα και έτσι υποσκάπτουν τις δυνατότητες ε, διαχείρισης ε, της αλληλευτικής ικανότητας. Επίσης, έχουμε δει αύξηση του στόλου. Βλέπουμε λοιπόν αύξηση της αλληλευτικής ικανότητας, της αλληλευτικής προσπάθειας με γρήγορη και άλλης αλληλείας από τις αρχές της δεκαετίας του 90 είδαμε μέση αύξηση αριθμού σκαφών γρηγρή στον δυτικό και κεντρικό ειρηνικό 3 με 5% το χρόνο. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 100 σκάφη είχαμε στις αρχές της ε, δεκαετίας του 90, ενώ τώρα έχουμε σχεδόν 350 σκάφη γρηγρή στην περιοχή αυτή όσον αφορά τις ε, τεχνολογικές πρόοδους, όσον αφορά τις σημαδούρες που συνδέονται με τα FADS, ο Ινδικός Ωκεανός αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα. Ξεκινήσαμε με ε, κάποιες ε, σημαδούρες, πλωτήρες ε, που είχαν περιορισμένο ε, φάσμα, περιορισμένο εύρος Όσον αφορά λοιπόν ε, τις ε, ηλεκτρονικές ε, συσκευές στο σκάφος, αναπτύχθηκε μια δεύτερη γενιά που ήταν πιο αποτελεσματικά και κατόπιν. Είχαμε την εφαρμογή συστήματος GPS στα σκάφη, έτσι λοιπόν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δορυφορικό σύστημα και τώρα πια έχουμε τέτοιους πλωτήρες με πολλές ε, συχνότητες ε, και έτσι λοιπόν ο Αλίας μπορεί εύκολα να διαπιστώσει αν αξίζει τον κόπο ή όχι να ε, πάει να δει τι γίνεται κάτω από ένα συγκεκριμένο φαντ. Μπορούν οι συσκευές αυτές να εντοπίσουν και το είδος και το μέγεθος των ψαριών. Ας συζητήσουμε λίγο τους δείκτες που έχουμε στις βάσεις δεδομένων των περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας. Η αλληλεία τροπικών θηνοειδών ε, στους ωκεανούς ε, του κόσμου ε, έχει φτάσει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Το 60% πρόσφατα αλλιεύθηκε από γρηγρή και σχεδόν το 65% της αλληλείας με γρηγρή σε όλο τον κόσμο έχει γίνει με βάση τέτοιες πλωτές διατάξεις. Είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση ανάμεσα στα φάντε και τα φυσικά απλωτά αντικείμενα. το free school fishing είναι η αλληλεία ε, κοπαδιών ε, τόνου που ε, απλά κολυμπάνε ελεύθερα, δεν έχουν συγκεντρωθεί από μια τέτοια διάταξη. Από τη δεκαετία του 90 η αλληλεία τόνου με γρηγρή έχει αυξηθεί κατά 60%, 33% στην αλληλεία ελεύθερων κοπαδιών, ενώ η αύξηση αλληλεία σε, σε πλωτά αντικείμενα ε, έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 82%. Και γενικά αντικατοπτρίζουμε εδώ τα μοτίβα αλληλείας ε, στον δυτικό κεντρικό ειρηνικό. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις ε, τα μοτίβα αλληλείας να διαφέρουν κάπως από τα μοτίβα στον κεντρικό ειρηνικό. Εδώ βλέπετε τέσσερα διαγράμματα. Την εξέλιξη θηνοειδών από τη δεκαετία του 60 και μετά. Ε, πάνω αριστερά βλέπετε συνδυασμό των τριών ε, ε, ειδών. Πάνω δεξιά βλέπετε τον κυτρινόπτερο τόνο που πρόσφατα είχαμε μείωση. Μην ξεχνάτε ότι αλλιεύεται και με παραγάδι και με γρηγρή καθώς και με άλλα είδη αλίας. Ε, το ίδιο ισχύει για τον μεγαλόφθαλμο τόνο, κάτω αριστερά. Στη περίπτωση της παλαμίδας όμως, που γενικά αλλιεύεται κυρίως με γρηγρή, ιδιαίτερα στον ε, δυτικό ειρηνικό βλέπετε συνεχή αύξηση και η αλληλεία με διατάξει κέντρου συχθείων ε, στόχο ακριβώς έχει να διατηρήσει τα επίπεδα αλληλεία ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετία του 90 και μετά. Εδώ βλέπετε την ε, συνολική αύξηση στα, στην αλληλεία μέχρι γρηγρή. Αριστερά βλέπετε την ε, ελεύθερη αλληλεία χωρίς δηλαδή πλοκά αντικείμενα. Βλέπετε κάποια αύξηση. Αριστερά βλέπουμε πολύ μικρό ποσοστό μεγαλόφθαλμου τόνου. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή στο κάτω μέρος του διαγράμματος, ενώ δεξιά βλέπουμε ε, μεγαλύτερο ποσοστό μεγαλόφθαλμου τόνου. Βλέπετε όμως ότι η αλία παλαμίδας ε, κυρίως ε, αντιπροσωπεύει την αύξηση που βλέπουμε. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί με αύξηση της αλλιευτικής προσπάθειας, αύξηση του αριθμού ή και αύξηση της δυνατότητας αλίας, αλευτικής ικανότητας. Ε, αλλά δεδομένων αυτά που γνωρίζουμε, μάλλον ε, δεν ισχύει το ότι υπάρχει μεγαλύτερο αριθμό ψαριών. Όσον αφορά τις τάσει ε, στις αναλογίες, ε, για, ε, ε, τις αναλογίες αλλιευμάτων για τα γρήγρη, βλέπετε ότι υπάρχει αύξηση 1% το χρόνο στο διάγραμμα πάνω από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Η γκρίζα γραμμή είναι η παλαμίδα. Βλέπετε πάλι ανάλογα μεγέθη αύξησης κάτω. Βλέπετε ε, σε τροπικές περιοχές με FAD. Εδώ δεν είναι πολύ καθαρή η εξέλιξη. Βλέπουμε ότι η παλαμίδα σε όλο τον κόσμο ε, αλλιεύεται κατά 65% από φάντε, ενώ τα τροπικά είδη ε, εδώ βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Α κοιτάξουμε λοιπόν τις δείκτες ε, αλλιευτικές προσπάθειε που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων των περιφερειακών ε, οργανώσεων αλληλείας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε εδώ κάποιε περιπτώσεις όπου δεν είχαμε αλίευμα και όπου είχαμε στην αλλιευτική προσπάθεια με ε, γρηγρή. Από τη δεκαετία του 90 η αλλιευτική προσπάθεια με γρηγρή έχει αυξηθεί περίπου κατά 2% το χρόνο. Η αύξηση της ε, αλίας γρηγρή με κάποιο αντικείμενο πλωτό έχει αυξηθεί κατά 70% διότι ξεκίνησε και από πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τη ελεύθερη αλλιεία. Βλέπουμε ότι η αλία κοντά σε πλωτά αντικείμενα είναι κατά 50% πιο παραγωγική από ότι η ελεύθερη αλία, αλλά στην περίπτωση του κυτρινόπτερου ε, τόνου δεν ε, βλέπουμε να προκύπτει αυτό το μοτίβο. Εδώ βλέπουμε ότι η αλληλεία κοντά σε πλωτά αντικείμενα και η ελεύθερη αλληλεία είναι περίπου η ίδια. Στην περίπτωση του μεγαλόφθαλμου η αλία κοντά σε πλωτά αντικείμενα ε, ε, είναι δεκαπλάσια από την ελεύθερη αλία. Εδώ βλέπετε την τάση για την αλλιευτική προσπάθεια με διατάξει συγκέντρωση ηχθείων ε, και με την ελεύθερη αλία. Βλέπετε ότι η αύξηση ήταν περίπου ίδια και για τα δύο είδη αλίας, όπως είπα όμως οι διατάξει συγκέντρωση ηχθείων βρισκόντουσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις αρχές τη της ε, του 90 από τη ελεύθερη αλληλεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι η γενική αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη για τις ε, διατάξει συγκέντρωσης ηχθείων από ότι για την ελεύθερη αλληλεία. Πάντως ε, γενικά τα νούμερα είναι περίπου τα ίδια για τα δύο αυτά είδη αλληλεία. Θα πρέπει και πάλι να πω ότι ε, αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιοχές. Ε, στον ε, Ατλαντικό έχουμε περισσότερη ελεύθερη και στον Ινδικό ωκεανό, κυρίως στην δυτική στο, στον δυτικό κεντρικό ειρηνικό έχουμε τις εξελίξεις αυτές. Βλέπετε εδώ πέρα την σχετική αποτελεσματικότητα των διατάξεων συγκέντρωσης ηχθείων και των άλλων διατάξεων. βλέπετε ότι ο μεγαλόφθαλμος τόνος ε, αλλιεύεται, ότι η αλλία ε, μεγαλόφθαλμου τόνου κοντά σε πλωτά αντικείμενα είναι η δεκαπλάσια από ό,τι κατά τα άλλα. Ε, βλέπετε η παλαμίδα που είναι η πορτοκαλιά γραμμή πάνω-πάνω, έχουμε την διπλάσια ποσότητα. Και μετά έχετε τα τροπικά θηνοειδή γενικά που είναι η γκρίζα γραμμή και εδώ η διαφορά είναι περίπου 50%. ενώ για τον Κιτρινόπτερο βλέπουμε ότι ο μέσος όρος είναι περίπου ένα, το οποίο σημαίνει ότι ε, η διαφορά είναι ελάχιστη. Επίσης, ε, με την πρόοδο της τεχνολογίας, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πλωτήρες, έχουμε δει αύξηση των επιτυχών αληφτικών ταξιδιών ανά ημέρα. Βλέπετε, η, κίτρινη, η πράσινη γραμμή είναι για τον Ινδικό ωκεανό και έχουμε στοιχεία και για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι για άλλους στόλους. Η πράσινη γραμμή αριστερά ε, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση όσον αφορά τον μέσο αριθμό ε, αλληλευτικών ταξιδιών ανά ημέρα. Ενώ δεξιά στον Ινδικό ωκεανό βλέπουμε ότι επίσης υπάρχει αύξηση υπάρχει κάποια διακύμανση, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η αλληλεία με φάτζ είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι η ελεύθερη αλληλεία. Να αναφερθώ τώρα στον στόλο και τους δείκτες σχετικά με το πόσα φάντα έχουμε στον ωκεανό. Το 2013 τα γρηγρεί σε όλο τον κόσμο, μεγάλης κλίμακας, ε, μάλλον ανέρχονται σε 700 σκάφη. Ε, αυτά τα στοιχεία τα έχουμε συνδυάζοντας στους καταλόγους ε, των διαφόρων περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας. Ξέρουμε τον αριθμό των σκαφών ε, που έχουν καταχωρηθεί, αλλά μερικά μπορούν να αλλιεύουν σε πάνω από μία θάλασσα, σε πάνω από έναν ωκεανό. Επίσης υπάρχουν σκάφη στους καταλόγους αυτούς που τελικά δεν αλλιεύουν. Αλλά γενικά φαίνεται ότι το 75% των σκαφών αυτών αλλιεύουν ένεργα στους ωκεανούς του κόσμου. Υπάρχει και κάποια δυσκολία όσον αφορά την καταμέτρηση των φάτ που χρησιμοποιούνται το κάθε χρόνο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ένα σύστημα παρακολούθησης που να μας επιτρέψει αυτή την ε, ανείχνευση των ΦΑΤ σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 13.000 ε, σταθερά ΦΑΤ ε, που υποστηρίζουν περίπου 8.000 σκάφη που αλλιεύουν τόνο και θηνοειδή. Όπως σας είπα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός, πολλά από αυτά όμως βρίσκονται στη Μεσόγειο και δεν χρησιμοποιούνται για την αλληλεία τόνου. Υπολογίζουμε ότι τα ε, ελεύθερα φαντ ε, ανέρχονται σε 91.000 το χρόνο. Μια προηγούμενη μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από τους παραγωγούς. Βλέπετε εδώ διάγραμμα ανά σημαία και ανά κατηγορία σκάφους. Ε, θεωρούμε ότι ε, το σκάφος με χωρητικότητα πάνω από 335 κυβικά μέτρα θεωρείται μεγάλο σκάφος, ενώ οτιδήποτε πιο μικρό από αυτό θεωρείται μικρό σκάφος, όπως βλέπετε. Έξι ή δέκα 5 ή 10 χώρες ε, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεξιά. Βλέπετε... Συγγνώμη, δεξιά βλέπετε τον αριθμό των ε, σκαφών και αριστερά βλέπετε ε, τον κυβισμό, τη χωρητικότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό σκαφών βρίσκεται στον ε, κεντρικό, ανατολικό, ε, κεντρικό και δυτικό ειρηνικό. Τα σταθερά FAD. Για τα σταθερά φάντα, τα στοιχεία αυτά ε, προέρχονται από επιρογνώμονες χρησιμοποιούνται κυρίως ε, για να αλλιευθούν ε, τόνοι και σχετικά είδη. Τα περισσότερα από αυτά τα φατ βρίσκονται στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες ε, και Παππούα Νέα Γουινέα που αντιπροσωπεύουν το 85% αυτού του είδους των φατ. Το 95% τα 100 βρίσκεται στον κεντρικό και δυτικό ειρηνικό. Όσον αφορά τα παρασυρώμενα φάτζ, υπολογίζουμε ότι χρησιμοποιούνται 91.000 το χρόνο. Πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στον κεντρικό και κεντρικό δυτικό ειρηνικό και ακολουθείται η περιοχή αυτή από τον ανατολικό ειρηνικό κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων τροπικού τόνου. Έχουμε 13 τέτοια αποθέματα τα οποία καταγράφουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν ε, συμπεριλαμβάνω εδώ την... Ε, συμπεριλαμβάνουμε εδώ την ε, Παλαμίδα. εκτός από τον κυτρινόπτερο στον Ατλαντικό και, στην, ε, και στον Ανατολικό Ειρηνικό, είδαμε ότι βρίσκονται σε καλά επίπεδα όλα αυτά τα αποθέματα. Ε, και μάλιστα με επίπεδα βιομάσας που θα μπορούσαν ε, να οδηγήσουν στην μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Στην τρίτη στήλη βλέπετε το ποσοστό παρεπιπτών των αλλιευμάτων. Όπως αυτό αντικατοπτρίζεται ε, στις πληροφορίες ε, της ε, Επιστημονικής Επιτροπής ISFF. όσον αφορά την εκμετάλλευση των αλλιευμάτων αυτών, όλα τα αποθέματα παλαμίδας με βάση τις ε, πιο σύγχρονες εκτιμήσεις ε, βλέπουμε ότι ε, έχουν χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας και θα προσέξετε ότι ο μεγαλόφθαλμος τόνος και ο κιτρινόπτερος έχουν ποσοστά θνησιμότητας πάνω από αυτά που μπορούν να οδηγήσουν σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν μέτρα διαχείρισης που υπολογίζεται ότι θα μετριάσουν αυτά τα ποσοστά θνησιμότητας και θα μπορέσουμε έτσι να οδηγηθούμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Με εξαίρεση τον ε, ε, Δυτικό Κεντρικό Ειρηνικό. να συνοψίσω τις πληροφορίες. Το 93% ε, των αλλιευμάτων ε, τροπικού τόνου προέρχεται από υγιή αποθέματα και μεγάλο ποσοστό προέρχεται από αλλία που χρησιμοποιεί φάτς και αυτό κυρίως οφείλεται στην παλαμίδα. Η χρήση των ΦΑΤ δεν οδηγεί απαραίτητο σε υπεραλίευση, σε υπερβολική εκμετάλλευση δηλαδή αν και η αλίευση μεγάλων ε, όγκων ε, μικρών τόνων, δηλαδή του μεγαλόφθαλμου του κοιτρινόπτερου, μπορεί να οδηγήσουν ε, σε μπορούν να μειώσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Γενικά, είπαμε, τα αποθέματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά η αύξηση της πίεσης από την αλία μπορεί να αλλάξει αυτά τα δεδομένα και αν συνεχιστεί η αλία με φαντ ε, στον ε, ρυθμό που είδαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό θα αυξήσει την ε, πίεση για τα αποθέματα αυτά, εκτός εάν αντισταθμιστεί από μείωση σε άλλα είδη αλίας ή αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που θα μετριάσουν την κατάσταση, που θα μετριάσουν τις συνέπειες. Επίσης, Έχουμε το θέμα των ε, παρεπιπτών των αλλιευμάτων. Ε, μπορεί η αλληλεία με φάτ να έχει αρνητικές ε, συνέπειες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται μέτρα για να αποφευθεί αυτό. Όσον αφορά την χωρητικότητα, υπολογίζεται Ε, ότι τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα ε, ανέρχονται στο 2% των ε, στοχευμένων αλλιευμάτων τόνου. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την περιοχή, μπορούν να φτάσουν μέχρι 8% στον Ατλαντικό. Υπάρχουν όμως κάποιες βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί για τη χρήση των γρηγρή με φατ και έχουν μεταφερθεί στους εφοπλιστές και ιδιοκτήτες πλοίων σε όλο τον κόσμο. και επίσης έχουν γίνει έρευνες σε συνεργασία με αλληλείς. Αυτό συνεχίζεται. Εξερευνούνται οι τεχνικές που μπορούν να μετριάσουν τα, τις αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τα παρεπίπτωτα λιεύματα. δεξιά μια ε, υπόθεση ότι υπάρχουν ε, κάποιοι οδηγοί με τέτοιες ε, καλές Όσον αφορά τους καρχαρίε και τι θαλάσσιες χελώνες. Οι θαλάσσιες χελώνες ε, είναι γνωστό ότι αποτελούν παρεπίπτον αλίευμα στην αλία με φάτο, παρότι ο αριθμός ε, των ε, χελώνων που πεθαίνει στα γρηγρή τώρα πια είναι πολύ μικρότερος από ότι με άλλα είδη εξοπλισμού όπως είναι τα παραγάδια. Επίσης έχουμε τους καρχαρίες, τον μακροπτέρυγο καρχαρία και τον λίο καρχαρία φαίνεται ε, ότι η αλείς αυτή στους, στους καφέδες αυτούς μειώνεται ο αριθμός τα τελευταία χρόνια. Μία από τις καλύτερες πρακτικές για να μειώσουμε το πρόβλημα θα ήταν η χρήση FAD ε, όπου να μην υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτούν στα δίχτυα καρχαρίες, ενώ ε, επίσης σε μια καλή πρακτική είναι να απελευθερώνονται ζωντανά τα ζώα αυτά στο σκάφος. Ενώ άλλη, εναλλαγή, ε, άλλη εναλλακτική λύση είναι να υπάρχουν τρόποι να απελευθερώνονται κατευθείαν από τα δίκτυα. Υπάρχουν ε, κάποια πειράματα που γίνονται αυτή τη στιγμή με ε, πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Όσον αφορά τα παρεπίπτωτα αλλιεύματα άλλων ψαριών, ε, έχουμε πάνω από 15 τέτοια είδη, για παράδειγμα τα ψάρια ιστιοφόρος, κομίτης, βαλίστρες κλπ. Αυτά λοιπόν ε, τα ψάρια αλλιεύονται ως παρεπίπτον αλλιεύμα στην περίπτωση αλλιείας ε, ε, της παλαμίδας του κυτρινοπτέρου και του ε, μεγαλόφθαλμου τόνου. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ πέρα είναι τα απόβλητα. Τα περισσότερα ψάρια που αλλιεύονται με γρηγρή απορρίπτονται στη θάλασσα παρότι σημειώνω ότι τουλάχιστον στον Ανατολικό Ατλαντικό έχει αναπτυχθεί μια αρκετά καλή αγορά για αυτά τα κατά τα άλλα ανεπιθύμητα είδη. Υπάρχουν ε, ψάρια τα οποία πολλούνται στις ε, χώρες της Δυτικής Αφρικής που κατά τα άλλα είναι ανεπιθύμητα. Υπάρχει λοιπόν ε, η ιδέα διατήρησης των παρεμπιπτών των αλλιευμάτων για να λυθεί το πρόβλημα των αποβλήτων, των απορρίψεων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί εάν ε, δεν αλλιεύει κανείς ε, μικρά κοπάδια τόνου, διότι εκεί συνήθως το ποσοστό άλλων ψαριών είναι μεγαλύτερο. Μια σειρά συστάσεων που θέλαμε να παρουσιάσουμε είναι η εξή Πρώτον, ε, να αποφύγουμε περαιτέρω ε, πίεση στα αποθέματα των ε, τροπικού τόνου με περαιτέρω αύξηση των ΦΑΤ χωρίς αντισταθμιστικές μειώσεις σε άλλα είδη αλίας. Δεύτερον, να εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης της κινητοποίησης και χρήσης των ΦΑΤ μέσω των περιφερειακών οργανώσεων αλίας. Τρίτον, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ε, που να επιτρέπει την παρακολούθηση της ε, απόδοσης των σκαφών επίσης ε, να να ελαχιστοποιηθούν τα περιπίπτωτα αλλιεύματα με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών όπως αυτές που ήδη αναφέραμε και που ήδη έχουν εντοπιστεί με την συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλλιέων και επίσης να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Πέμπτον, να παρακολουθούν τα παρεπίπτουν τα αλλιεύματα και να ε, επαληθεύεται η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών ε, με είτε ανθρώπινους παρατηρητές είτε με ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης ή και με τα δύο. Ε, η πλήρης παρακολούθηση της αλίας γρηγρή με φαντ θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των παρεμπιπτών αλληλευμάτων. Και τέλος, θα πρέπει να παρέχονται δεδομένα μέσω των ε, περιφερειακών ε, οργανώσεων αλληλείας ε, για να παρακολουθείτε η αύξηση της αλληλευτικής προσπάθειας. Και επίσης να χρησιμοποιείτε και το, σύστημα, το, σύστημα παρακολουθήσης των σκαφών. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την βοήθεια που μου παρήχαν διάφοροι άνθρωποι και συνάδελφοι ε, πάντως οι απόψεις που ε, παρουσιάζω όπως και οποιοδήποτε λάθος ε, μπορεί να έχει γίνει είναι αποκλειστικά δικό μου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Σκότ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, κυρία Φράγα, κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ τον δόκτωρα Σκότ για αυτή την έκθεση και για την παρουσίασή της. Είναι πολύ αντικειμενική αυτή η έκθεση. Ε, αναλύει τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΦΑΤ. Θέλω όμως να υπογραμμίσω κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στις συστάσεις. Ξέρω ότι είναι εμπειρογνώμονας, έχει εργαστεί σε πολλές περιφερειακές οργανώσεις ε, Να σας ρωτήσω λοιπόν το εξή. Λέτε, πολύ σωστά, ότι το σημαντικό είναι ο έλεγχος και η διαχείριση των ΦΑΤΣ στην Αλία. Και ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα, οι περιφερειακές οργανώσεις Αλίας. Ο κοινοτικό τόλος εμένα προσωπικά δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι ακολουθεί ένα κωδικά καλών πρακτικών, έχει εισάγει, εισάγει αυτή τη στιγμή σημαντικές ε, ε τεχνολογικές, ε, τεχνολογίες εχμής μάλλον. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ποιες ε, περιφερειακές οργανώσεις ε, αλίας γίνεται καλή δουλειά και μπορούμε να προχωρήσουμε. Στον δυτικό και κεντρικό ειρηνικό, για παράδειγμα, ε, ξέρουμε ότι είναι, γίνεται μεγαλύτερη χρήση των FAD. Εκεί ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και ο λιγότερος έλεγχος. Θα μπορούσατε να μας δώσετε όμως λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. για να δούμε πώς λειτουργούν οι περιφερειακές οργανώσεις ε, διαχείρισης αλληλείας, η πόδα. Ευχαριστώ πολύ, ο κ. Ζωμέβα. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Ακόμα μία φορά, κύριε Σκότ. Παρόμοια ερώτηση έχω με την ερώτηση της κυρίας Φράγκα, που αφορά το θέμα της διαχείρισης. Το σαφές μετά την ανάγνωση της έκθεσής σας και την παρουσίασή σας είναι ότι έχουμε την εξής κατάσταση. Είμαστε πολύ μακριά από τη φάση της διαχείρισης και το πολύ πολύ να εξασφαλίσουμε κάποιους εθελοντικούς τρόπους ή τους ατομικούς τρόπους με τους οποίους μειώνονται τα παραλιεύματα, τα παρεμπιπτόντα Δεν υπάρχουν λοιπόν κανόνες. Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες ελέγχου. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Για να δώσω έμφαση σε κάποια στοιχεία της παρουσίασής σας και να διευρύνω μάλιστα και το πλαίσιό της. Καταρχάς, η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Έχουμε μειωμένες αποδόσεις τώρα. Τι επίπτωση μπορεί να έχει στα αποθέματα μεγάλου οφθαλμού τόνου. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεύτερο ερώτημα. Διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, ειδικά για τον τόνο που αλληλεύεται σε τροπικά κλίματα. Ο χρόνος αναζήτησης του τόνου δεν συνυπολογίζεται για να λάβουμε υπόψη την επίπτωση που έχουν τα φαντ στα αλλιεύματα. Οι εναλλακτικοί δείκτες ε, αλληλευτικής προσπάθειας σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμοι για να κάνουμε αξιολόγηση της κατάστασης των αποθεμάτων. Μία διευκρινιστική ερώτηση. Δεν έχει κανένα ίχνος επίκρισης αυτή η ερώτηση. Πηδάω τώρα από το ένα στο άλλο θέμα, το ξέρω. Αλλά το τρίτο είναι ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Κάτι που ανέφερατε στις στάσεις στο τέλος. Οι, μακροπρόθεσ... οι μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις αν δεν αλλάξει τίποτα. Έτσι, οι μακροπρόθεσμες πάντα. Εάν αυξηθεί η χρήση των φαντς. Ξέροντας ότι πιάνουμε μεγάλα ποσότητα, μεγάλες ποσότητες νεογνών. Ποια θα είναι η επίπτωση στη βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης σε αυτό το επίπεδο, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν και κάτι συναφές. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα των ποσοστών θνησιμότητας. Για να δω πού το πάμε, πού θα καταλήξουμε αν δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ. που ήρθατε. Δυστυχώς δεν άκουσα το πρώτο τμήμα της παρουσίασής σας. Ζητώ συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να, προσπάθησα να διατρέξω την έκθεση. Και έχω την αίσθηση ότι οι συστάσεις που αναφέρεται στο τέλος του κειμένου είναι πολύ σοβαρές. Καταρχάς να μην αυξήσουμε την πίεση στα λιεύματα με περαιτέρω χρησιμοποίηση των ΦΑΤ χωρίς μείωση αλλού της προσπάθειας. Αν συνολικά αυξηθεί η αλλιευτική προσπάθεια θα υπάρξει πρόβλημα. Και επίσης ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, συστήματα παρακολούθησης ε, στα επίπεδα, σε όλα τα στις περιφερειακές οργανώσεις Υπάρχει πρόοδος, μια και είσαστε μέσω των περιφερειακών οργανώσεων αλίας για να αντιμετωπίσουμε εκεί, σε αυτό το επίπεδο, το θέμα των FADS. Γιατί Βασικά εστιάζουμε στη χωρητικότητα και στο μήκος των σκαφών, στην αλληλευτική προσπάθεια των σκαφών, αλλά ποτέ στο, στην ποσότητα των χρησιμοποιούμενων φαντ. Πόσα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται, πού, πότε. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το σημείο. Και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτή την κατεύθυνση. Για τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Πάντα με απασχολεί αυτό το θέμα. Τα παραλιεύματα δεν αφορούν μόνο άλλα είδη του τόνου. Δεν είναι μόνο, μόνο καρχαρίες και χελώνες, αλλά άλλα είδη ανεπιθύμητα τόνου. Είπατε ότι, περίπε, ότι μπορεί να είναι στον Ατλαντικό 2 με 8% αυτά τα παραλιεύματα. Μιλάμε 2 με 8% κατά βάρο. ή μιλάμε άλλα είδη πλην τόνου ή μιλάμε για νέο γνούς τόνου που δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να ψαρεύουμε με αυτά τα μέσα αλίευσης. Γιατί μιλάμε ακριβώς λοιπόν. Άλλος κανείς. Ο Τόμας έχει την, το λόγο, ο Τόμας Κότ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε διάφορα ερωτήματα με μία απάντηση. Υπάρχουν, ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν τη διαχείριση των ΦΑΔ και αν υπάρχουν σχέδια διαχείρισης των ΦΑΔ. Υπάρχει πρόοδος στις περιφερειακές οργανώσεις αλληλεία σε σχέση με τα ΦΑΔ, αλλά είμαστε ακόμα στην απαρχή. Στον IOTC και στον ITTC υπάρχουν σχέδια για συλλογή δεδομένων Με την εξαίρεση του ITTC όμως, ε, τα δεδομένα αυτά ακόμα δεν τα έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, στην Ευρώπη, η απέτηση για παρακολούθηση και καταγραφή της χρήσης των FAD και τα σχέδια ανάπτυξης και χρησιμοποίησης των FAD ε, βασικά αντιγράφουν αυτά που έχει κάνει ο IOTC και ο ITTC. Στο κεντρικό και δυτικό ειρηνικό δεν υπάρχουν ακόμα συμπεφωνημένα σχέδια διαχείρισης των ΦΑΝΤ. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, θα πρέπει να εστιάσουμε σε μια συμφωνία. Φτάσαμε κοντά στη συμφωνία, αλλά δεν τα καταφέραμε σε διάφορες περιοχές, από ό,τι ξέρω. Ένα άλλο ερώτημα που ακούστηκε αφορούσε τους κανόνες για τη διαχείριση των ΦΑΝΤ. Πώς ε, θα προσμετρήσουμε την επίπτωση με καλύτερο τρόπο της αλίευσης με ΦΑΝΤ. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε καταρχάς λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα ΦΑΝΤ, πού χρησιμοποιούνται και μόνο από αυτά τα αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να φτιάξουμε σχέδια διαχείρισης. Μπορούμε και μέσω της συνεργασίας με τους γεωργούς να συλλέξουμε δεδομένα βέβαια, πέρα από τα σχέδια διαχείρισης. Προηγουμένως μίλησα για πρόσβαση σε λεπτομερείς ε, πληροφορίες για τη θέση των σκαφών, ε, των ΦΑΔ και δεδομένα από τους από τις ηχοεντοπιστικές συσκευές ε, και τα σόναρ. Υπάρχουν κάποιες γενικές συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε κοινέ αναλύσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν για να δούμε πώς είναι η τεχνολογική επίπτωση ε, στην ικανότητά μας να ψαρεύουμε περισσότερα ψάρια. Ε, το να έχουμε πρόσβαση στις, ε, στα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ένα άλλο ερώτημα που ακούστηκε αφορά την ε, μειούμενη απόδοση. Η στον ε, μεγαλόφθαλμο και κυτρινόπτερο τόνο. Αυτοί οι δύο τόνοι ψαρεύονται με διάφορους τρόπους, ε, όχι μόνο με γρήγορη με σειρώμενη, σειρώμενα δίχτυα, όπως είναι περίπτωση της, ε, της Παλαμίδας. Και φυσικά οι νεογνοί του μεγαλόφθαλμου, ας πούμε, έχουν ε, μειωθεί. Ε, είναι μικρότεροι από ό,τι, ας πούμε, του, της παλαμίδας. Γιατί, πώς γίνεται αυτό, ε, ψαρεύοντας πολλά ενήλικα ή πολλά νεογνά. Αν ψαρέψατε τα ενήλικα, γίνεται αμέσως. Αν ε, ψαρέψατε τα νεογνά, γίνεται αργότερα αυτή η συμπίεση. Η συνολική αλληλευτική πίεση επηρεάζει την κατάσταση των αποθεμάτων, συνολικά όμως. Τώρα, θέλουμε καταρχά μικρά ψάρια, ψάρι να ψαρεύουμε ή μεγάλα ψάρια. Εξαρτάται από τις αγορές που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Παραδείγματο χάρη την βιομηχανία κονσέρβας. Αυτά θέλουν μικρο... Αυτή η μεγαλα ψαρια εξαρταται απο τι αγορες θέλει την βιομηχανια κονσερβας μικρο ψάρι ε, σε σχέση με τη βιομηχανία φρέσκου ψαριού, όπου θέλει μεγαλύτερο ψάρι. Δεν μπορώ να ρυθμίσω αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις πολιτικές που έχουμε για τις αγορές και τις πολιτικές που έχει η εκάστοτε χώρα. Δεν συμφωνούν ποτέ όλες οι χώρες επί μίας πολιτικής. Πάντα θα γίνει διαπραγμάτευση. Είναι θέμα δούνε και λαδίν. Αυτό κάνει την άποψή μου. Για τη διαχείριση της προσπάθειας και τις μονάδες ε, για την προσμέτρησή της. Ε, γίνεται μια συζήτηση. Είναι ένα θέμα που επηρεάζεται πολύ από την τεχνολογία. Έχουμε 23 παράγοντες εντοπίσει που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του γρηγρή. Παραδείγματος χάρη, βοηθητικά σκάφη, ελικόπτερα, το να βάζουμε ε, πλωτήρες στα, φέτζ, στα φάντζ. Είναι δύσκολο να τα διαχωρίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, να δούμε το καθένα πώς επηρεάζει ας πούμε τελικά, πόσο αποτελεσματικό είναι το κάθε αλληλευτικό εργαλείο στην αλληλεύση του κάθε είδους. Στις στατιστικές δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να δούμε αυτές οι τεχνολογίες, αυτές οι συσκευές, πώς επηρεάζουν τα αλληλεύματα. Επιλέξαμε λοιπόν εδώ στην παρουσίαση να σας μιλήσουμε για τον αριθμό των εργαλείων και των συσκευών αυτών. Θετικές ύπαρξη συσκευών ή μη ύπαρξη, πούμε, συσκευών. Είναι μια χοντροειδής αντιμετώπιση, πιο προσεγγιστική, αλλά αυτή χρησιμοποίησαμε εδώ. Για την αξιολόγηση των αποθεμάτων χρησιμοποιούμε παρόμοια είδη μέτρων, μερικές φορές Πάσουμε και κάποιες υποθέσεις. Γιατί δεν μπορούμε πραγματικά να ξέρουμε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές. Τι επιπτώσεις θα έχουν, ας πούμε, σύντο χρόνο. Στον Ατλαντικό μερικές φορές λέμε ότι έχουμε μια αύξηση, ας πούμε, 3% ε, το χρόνο ε, στα γρηγρή. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση. Ξέρω ότι δεν είναι η πιο ακριβής. Γιατί αυτές οι τεχνολογικές, τα τεχνολογικά κέρδη δεν, γίνονται, δεν είναι σταθερά συν το χρόνο. Έχουμε αυξομοιώσεις. Μερικές φορές, ας πούμε, έχουμε ξαφνική αύξηση, ας πούμε, και μετά σταθεροποίηση, μείωση κτλ. Χρειαζόμαστε πιο λεπτομερή, όπως σας είπα, επιχειρησιακά στοιχεία. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ηλεκτρονική παρατήρηση που έχουμε ε, πάνω στα γρηγρή. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα από ηλεκτρονικά μέσα πάνω στα γρηγρή ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε την επίπτωση που έχει κάθε τεχνολογική εξέλιξη και συσκευή. Αυτή ήταν μία από τις συστάσεις, ήταν λίγο σκοτεινή, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα και τα στοιχεία που έχουμε από αυτά. Είναι πολύ σημαντικό για να αξιολογήσουμε την κατάσταση των αποθεμάτων. Επίσης, μακροπρόθεσμα, τι γίνεται. Προσπάθησα να το πω ότι γενικά Έχουμε μεγαλύτερη αλληλευτική προσπάθεια, αυξάνεται ο ρυθμό των σκαφών ε, και δεν είναι μια κατάσταση που έγινε ξαφνικά. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Υπάρχουν ε, σχέδια διαχείρισης στον ε, Ινδικό και στον Ειρηνικό, λίγο λιγότερο στον Ατλαντικό και στον Ανατολικό Ειρηνικό. Και αυτά τα πράγματα επηρεάζουν την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα σκάφη στον δυτικό ας πούμε, ειρηνικό αυξάνονται. Αυξήθηκαν μάλλον από 100 στα 300 σκάφη τα τελευταία 25 χρόνια. Επομένως, τεράστια αύξηση. Πολλά κέρδη ε, στα λιεύματα. Επομένως, δεν είναι μόνο το γρήγορο ότι χρησιμοποιείται, δεν είναι μόνο αυτή η μορφή αλίευσης. Υπάρχουν και άλλες μορφές ε, αλίευσης ε, μειώνεται ένα συγκεκριμένο απόθεμα, αλλά συνολικά έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα αποθέματα. Πρόκειται για ένα πακέτο. Δεν μπορώ να εστιάσω σε ένα στοιχείο και να ξεχάσω τα άλλα. Αν παραμείνει η αλίευση με παραγωδιάρικο όσο έχει σήμερα και μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε καλύτερες αποδόσεις από την αλίευση με παραγαδιάρικο, εάν μειωθούν άλλες μορφές αλίευσης. για αυτό το 2 με 8% κατά βάρος αύξηση. Το, το μετρήσαμε κατά βάρος, αν το μετρήσουμε κατά απόλυτες τιμές, προφανώς θα είναι διαφορετικό το ποσοστό. Σε τόνους όμως, τα νεογν... τα... οι νεογνοί ε... καρχαρίες και τα λοιπά, όλα τα είδη ε... τα συνυπολογίσαμε μέσα σε αυτό το ποσοστό 2 με 8%. οστεώδεις ηχθείες, όλα τα είδη υπολογίστηκαν σε αυτό το ποσοστό 2 με 8%. να Otra cuestión aclarada. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις όχι. Ε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοτ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Διάφορα. Δεν υπάρχει κάτι εδώ. Από τη δική μου πλευρά, θέλει κανείς να θέσει κάποιο θέμα στα διάφορα. Όχι. Ανακοινώσει του Προέδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν οι συντονιστές. Βλέπετε την ανακοίνωση, την έχετε στα χέρια σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, όχι. Επόμενη συνεδρία 18 Μαρτίου, 9 με 12 και μισή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.